είναι οι δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τη Σύνοδο κορυφή των G20 στο Πίτσμπουργκ που θα γίνει 24 και 25 Σεπτεμβρίου στο Πίτσμπουργκ. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτές τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής και θα δώσω πρώτα το λόγο στην ε, κυρία Σεσίλια Μάλμστρομ εκ μέρους του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε Αλμούνια. Μεγάλη χαρά για μένα που είμαι σήμερα εδώ για να εκπροσωπήσω τη Σουηδική Προεδρία η Προεδρία μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση Κορυφής G20 στο Pittsburgh στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και θα γίνει άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αύριο το απόγευμα, αύριο το βράδυ μάλλον, στις Βρυξέλλες για να προετοιμαστεί η κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως όλοι γνωρίζετε, η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική ε, κρίση ε, απέτησε να ληφθούν πάρα πολλά αντίμετρα. Χρειάστηκε Χρειάστηκαν πάρα πολύ ταχαία, μέτρα για να ελέγξουν την όλη κατάσταση. Μετά χρειάστηκε συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και αναπτύσσεται το G20 σαν ένας χώρος για συντονισμό, για τη λήψη μέτρων, για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Τα χρηματοσυντικά και νομισματικά μέτρα που θετήθηκαν πολύ γρήγορα ήταν απόλυτα αναγκαία, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε το χειρότερο κομμάτι της κρίσης. Η πλήρης υποστήριξη της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και φέτος και του χρόνου υπολογίζεται ότι είναι 5% του ΑΕΠ. Και οι κεντρικές τράπεζες έχουν βρει απαντήσεις για την κρίση, προσπάθησαν να κρατήσουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Οπότε έχουμε κάποια μικρή ελπίδα ότι περάσαμε τα χειρότερα όσον αφορά τα πολύ δύσκολα προβλήματα του χρηματοστικού τομέα. Αλλά η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να είναι ασταθής και ο κίνδυνος μιας επαναλήψεως της κρίσεως εξακολουθεί να εφίσταται. Ξέρουμε ότι η αύξηση της ανεργίας είναι ένα θέμα που θα κυριαρχεί ε, στην πολιτική ε, το επόμενο διάστημα. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αβέβαιη αλλά μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη. Ε, η συνεργασία και ο συντονισμός σε διεθνές επίπεδο θα είναι εξαιρετικά σημαντικά, θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια γενικότερη ανάκαμψη και θα ανοίξει ο δρόμος για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα βασίζεται στα στέρεα θεμέλια. Το G20 ε, ε, διαδραμάτισε και εξακολουθεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Οι G20 θα εξακολουθούν να συνεργάζονται με άλλου διεθνεί χρηματοστικού οργανισμού, την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, ώστε να υπάρχουν ε, επαρκεί πόροι και αποτελεσματική εσωτερική διοργάνωση, ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη και να εξασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα σε όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία των G20 οδήγησε και στα εξή σημαντικά αποτελέσματα. Καταρχά. Τώρα έχουμε μια κοινή ανάλυση των προβλημάτων τα οποία έπληξαν τις οικονομίες μας. Ίσως αυτό να μην ακούγεται σαν ένα μεγάλο βήμα πρόοδου, αλλά έχοντας μια κοινή άποψη για το χρηματοστικό σύστημα και τα οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν στην κρίση βοηθάει στη λήψη συντονισμένων αντίμετρων. Μετά πραγματοποιήθηκε μια πραγματική πρόοδο σε συγκεκριμένα μέτρα από τον οποίο είχαμε συμφωνήσει στην Οδοκορυφή στο Λονδίνο την περασμένη άνοιξη. Ε, γενικά πακέτα για την τόνωση των οικονομιών μα, η ενίσχυση του συντονισμού για την εποπτεία και τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών αγορών, παραδείγματι, δύο παραδείγματα. Ε, γενικότερα εξασφαλίσαμε το ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα έχει επαρκείς πόρους ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση για πιστώσεις και δεσμευτήκαμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τα διεθνή χρηματοστατικά ιδρύματα και τις δυνατότητες που έχουν να εποπτεύουν την παγκόσμια μακροοικονομική κατάσταση, ούτως ώστε αν παρόμοια προβλήματα ε, εμφανιστούν εκ νέου να μπορέσουν να μας προειδοποιήσουν έγκαιρα. Πολλά απομένουν να γίνουν, αλλά έχουμε σημειώσει μια σαφή πρόοδο, η οποία επετεύχθη μέσω συντονισμένων διεθνών μέτρων. Πιστεύω ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες του G20 κάναμε σημαντική πρόοδο σε βασικά θέματα που ήταν κάτι αναγκαίο για να βρούμε στατική απάντηση στην οικονομική και χρηματοπιστική κρίση. Συντονισμένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα σημαίνει ότι θα ηγείται η Ευρώπη και δεν θα ακολουθεί τα συζητούμενα και θα προσφέρει λύσεις που θα λαμβάνονται υπόψη όταν υιοθετούνται διάφορες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό ε, η Προεδρία κάλεσε του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων σε ένα δείπνο αύριο το βράδυ. Στόχο είναι να βασιστούμε στο πολύ επιτυχέ έργο του άτυπου γεύματο ε, ΕΚΟΦΗΝ και τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών των G20 στο Λονδίνο, τόσο ώστε να είμαστε έτοιμοι για τη Σύνοδο στο Πίτσμπουργκ. Ε, περιμένω ότι η αυριανή συνάντηση και η Σύνοδο στο Πίτσμπουργκ θα καλύψουν αυτά τα θέματα που προανέφερα σε γενικό πλαίσιο, αλλά έχουμε και άλλα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Ένα τομέα που πολλοί υπουργοί οικονομικών ε, εξετάζουν είναι το θέμα του ρόλου των συστήματος των, ε, των πόνους στο χρηματοσυντικό σύστημα. Υπάρχει συμφωνία μεταξύ Υπουργών Οικονομικών ότι θα πρέπει να ηγηθούμε, ούτω ώστε να έχουμε παγκόσμια πρότυπα και προδιαγραφές που θα είναι αποτελεσματικά, ούτως ώστε τα συστήματα αυτά των πόνους να μην ε, αποσταθεροποιούν την οικονομία και τα ποσά να είναι ανάλογα με τα επιτεύγματα. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της γενικότερη προσέγγισης για πιο ανοιχτή διαχείριση και μεγαλύτερη διαφάνεια στο χρηματοστικό τομέα, κάτι που είναι απαραίτητο για μελλοντική ε, σταθερότητα. Ε, ζητήθηκε από, το, από τον φορέα για τη σταθερότητα να μας δώσει κάποιες προτάσεις για συστήματα για αυτές τις αμοιβέ, για αυτά τα μπόνους. Ελπίζουμε να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα, πρακτικές στρατηγικές που θα μας εγγυώνται ότι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα θα δίνουν αμοιβέ και μπόνους τα οποία θα είναι σε υγιή επίπεδα και θα δίνονται με έθινο τρόπο. Ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία για την συνέχιση της τόνωσης των οικονομιών μας όσο αυτό είναι εφικτό και αναγκαίο. Επίσης θέλουμε αυτά τα μέτρα να καταργηθούν σταδιακά όταν δεν θα είναι πλέον αναγκαία. Να επιστρέψουμε σε ισολογισμένα δημοσιονομικά ε, όταν ε, επιστρέψουμε στη σταθερότητα. Ε, πρέπει να βρούμε στρατηγικέ διεξόδου. Έχει αρχίσει ο προβληματισμό μα αυτά και πιστεύω ότι ο συντονισμό και η μέθοδοι εφαρμογή αυτών των μέτρων θα είναι εξαιρετικά μεγάλη, εξαιρετική σημασία για να καταλήξουμε σε ισορροπημένη μακροπρόθεσμη ε, οικονομική ανάκαμψη. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό σαν πρόκληση και αντιμετωπίζουμε είναι η απασχόληση. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν θα αποφασίσουμε ποια μέτρα θα εφαρμόσουμε και χρειάζεται και σωστή διάδραση μεταξύ οικονομικής και διαθωτικής πολιτικής. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει ο προστατευτισμός να παραμείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, εκτός θα πρέπει να είναι ισότιμες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά. Αυτό είναι κάτι που απαιτεί σημαντικό συντονισμό όσον αφορά τον, ε, την εποπτεία του χρηματοστικού τομέα και τη ρύθμιση αυτού αλλά επίση και για την εξάλληψη των εκτάκτων μέτρων που υιοθετήθηκαν για την υποστήριξη του χρηματοστικού τομέα. Και θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε και σε διεθνέ επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Οι συζητήσει θα συνεχιστούν αύριο και στο Pittsburgh, αλλά και κατά το υπόλοιπο έτος περί μεταρρυθμίσεων για το διεθνή χρηματοστικά ιδρύματα. Θέλουμε να είναι ισχυρά τα ιδρύματα αυτά, θέλουμε να έχουν επαρκεί πόρου, θέλουμε να έχουν τη σωστή εντολή, ε, πολιτικούς και δομές διαχείρισης ε, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζεται και η δομή τους, τα μέλη τους. Αυτά τα θέματα είναι περίπλοκα και αλληλένδετα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα τόσο ώστε τα διεθνή χρηματοστικά ιδρύματα να συνεχίσουν το έργο τους που γίνεται όλο και πιο σημαντικό. Τέλος, ε, κυρίες και κύριοι, βεβαίως ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να λαμβάνονται με τρόπο οι πολιτικές αποφάσεις και στις συζητήσεις που δεξαχθούν για το κλίμα στην ε, Κοπενχάγη. Θέλουμε όλοι να δουν ότι θα έχουν τα σωστά κίνητρα για τη λήψη μέτρων, για τον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου και να έχουν τι σωστέ οικονομικέ στρατηγικέ για να υπάρχει μια εξέλιξη που θα είναι φιλική προ το περιβάλλον. Στόχο μα είναι η σύνοδο στο Πίτσπεργκ να οδηγήσει σε κάποιου προσανατολισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα πετύχουμε τα πάντα όσα θέλουμε να γίνουν σε αυτού του τομεί. Είναι περιπλοκότατα ζητήματα, αλλά υποσχόμεθα ότι η Προεδρία θα είναι πάρα πολύ υπεύθυνη στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάζει και θα υπερασπίζεται τη θέση Ευρωπαϊκή Ενώση. Και σε αυτό το πνεύμα προσβλέπω σε καρποφόρε συζητήσει με του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων αύριο το βράδυ και περιμένω συγκεκριμένα αποτελέσματα που άλλωστε αναμένει και ο κόσμο από τη Σύνοδο του Πίτσμπεργκ την επόμενη ε, εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε την προσοχή σα και προσβλέπω στο να ακούσω αυτά που έχουν να πούν τα μέλη. Thank you, madam. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσουμε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο Αλμούνια, Ζωακή Μαλμούνια να μας κάνει τη δήλωση εκ μέρους της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Μάλμστρομ, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Για πρώτη φορά λαμβάνω το λόγο εδώ στην Ολομέλεια με την καινούργια κοινοβουλευτική θητεία και θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ όλους σας για την εκλογή ή επανεκλογή σας. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι αισθανόμαστε ένα ε, βαθύτατο αίσθημα ευθύνης για να αντιμετωπίσουμε μία από τις μείζονε προκλήσεις της γενιάς μας που είναι η υπέρβαση αυτής της βαθύτατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης προκειμένου να επαναφέρουμε στους πολίτες μια εμπιστοσύνη, αισιοδοξία, να διαβρύνουμε το φάσμα των ευκαιριών και να επιτύχουμε ε, για όλους ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Τα θέματα που θα εξετάσουμε στη Σύνοδο Κορυφής του G20 στο Πίτσμπουργκ την επόμενη εβδομάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών μας. Πάντως έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι αυτό το θέμα θα μας απασχολήσει πολλάκις και στη διάρκεια της ε, κοινοβουλευτικής αυτής θητείας. Θα απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το θέμα αυτό των συνόδων κορυφής, ε, ε, αλλά και η συζήτηση των ε, διαφόρων πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα εξεταστούν εδώ διεξοδικά. Η Σύνοδος Κορυφής του Πίτσμπουργκ είναι η τρίτη που γίνεται σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων από τότε που ένα χρόνο και μία μέρα πριν κατέρευσε η Lehman Brothers και ξεκίνησε μία κρίση άνευ προηγουμένου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μετά τις πρώτες ε, διασκέψεις κορυφής ε, τον Νοέμβριο πέρυσι στη Ουάσιγκτον και το Λονδίνο φέτος τον Απρίλιο που έγιναν σε ε, επίπεδο κορυφής φάνηκε ότι το G20 διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο για το συντονισμό σε παγκόσμια κλίμακα της ανταπόκρισης σε αυτή την κρίση. Και η προσπάθεια για την ανέβρεση συντονισμένων λύσεων ήταν θεμελιώδης σημασία για να αποφευθεί μια βαθύτερη ύφεση αλλά και για να δημιουργηθούν τα θεμέλια ενός οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα αποτρέψει στο μέλλον την επανάληψη των ανισορροπιών και των υπερβολών που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε ε, πολύ αποφασιστικό ρόλο και στην πρώτη Σύνοδο Κορυφή ε, στη Ουάσιγκτον. Γιατί, όπω μα υπενθύμησε χθε ο πρόεδρο ε, Μπαρόζο, η πρώτη αυτή Σύνοδο Κορυφή ήταν Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία τη Γαλλική Προεδρία του Προέδρου Σαρκοζή ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέβαλε αποφασιστικά και στο προσδιορισμό των φιλόδοξων στόχων των δύο προηγούμενων συνόδων κορυφή και συμμετείχε ενεργά στην προπαρασκευή αυτών των συνόδων προκειμένου να καταλήξουμε όχι μόνο σε διακηρύξει επί της αρχής, αλλά σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και απτά αποτελέσματα. Για όλους τους Ευρωπαίους, τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να θεωρούνται ικανοποιητικά ως προς τη δράση τους. Επίσης, ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το βαθμό συντονισμού που επέδειξαν οι διάφοροι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο G20, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του G20 και που συμμετέχουν ε, ε, στην, ε, στο G20 ε, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησαν επάξια την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξέφρασαν τις κοινέ θέσεις όλων των χωρών μελών. Το Νοέμβριο η διάσκεψη κορυφής της Ουάσιγκτον συνέβαλε στο, οι, οι βασικές οικονομίες του πλανήτη που είναι απευθύνεται το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ να καταλήξουν σε ορισμένα σχέδια εναυσμάτων για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Πέρυσι το φθινόπωρο που υπήρξε μια κατάρρευση των πιστώσεων των, του παγκόσμιου εμπορίου και ένα τεράστιο οικονομικό σοκ που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2007 και επιταχύθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008. Λίγες μέρες μετά τη διάσκεψη κορυφής της Ουάσιγκτον πέρυσι τον Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης που το Δεκέμβριο έλαβε και την πολιτική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και αυτή ήταν η βάση της ευρωπαϊκής αντίδρασης ε, ως προς τις ε, δημοσιονομικές πολιτικές και τις πολιτικές ε, τόνωσης της ζήτησης. Σε συντονισμό με τα κράτη-μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Με βάση τις τελευταίες μας πληροφορίες, αυτά τα φορολογικά ενάβσματα που εφαρμόζονται σε προαιρετική βάση, αλλά και οι αυτόματοι σταθεροποιητέ, που είναι πολύ σημαντικοί δεδομένου του όγκου του φορολογικού μα συστήματο και του συστήματο κοινωνική προστασία, μα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι συμβάλλουμε στη ζήτηση ε, με τρόπο αντίστοιχο του 5,5% του ευρωπαϊκού PIB μεταξύ του 2009 και 2010. Και η Αμερικανική κυβέρνηση υιοθέτησε ένα σχέδιο ναυσμάτων πολύ σημαντικό. Βέβαια, οι αυτόματοι σταθεροποιητές στην Αμερική είναι χαμηλότεροι, οπότε ε, το άθροισμα των δύο αυτών μεθόδων μας οδηγούσε παρόμοιο αποτέλεσμα. Αλλά και χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, ο Καναδάς και άλλα μέλη του G20 υιοθέτησαν φορολογικά κίνητρα ε, και ενάβσματα παρόμοια με τα δικά μας. Στη διάσκεψη κορυφής του Απριλίου που έγινε φέτος, επιμείνουμε στην ταχύ εφαρμογή αυτών των σχεδίων των εναυσμάτων, στην εκτουσίνικης παρακολούθησή τους, αλλά και στην ανάγκη μετά από αξιολόγηση συμπλήρωσή τους. Σήμερα μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και τα φορολογικά αλλά και τα νομισματικά ενάψματα που υιοθέτησαν οι κεντρικές ε, τράπεζες αλλά και ε, τα ενάψματα που έδωσαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατάφεραν να συγκρατήσουν την ελεύθερη πτώση της οικονομίας, ώστε φέτος το φθινόπωρο να γινόμαστε μάρτυρες των πρώτων συμπτωμάτων της σταθεροποίησης. Όπως ακούσατε και στην παρουσίασή μου που έγινε πριν από δύο μέρες στις Βρυξέλλες. Και έτσι δεν χρειάστηκε με τα τελευταία στοιχεία να αναθεωρήσουμε προς το χειρότερο τις προηγούμενες μας προβλέψεις. Βέβαια, η οικονομική δραστηριότητα δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της αν καταργηθούν σήμερα τα ενάβσματα. Παρόμοια με τα κίνητρα αυτά και αν αφαιρεθούν αυτά τα κίνητρα, υπάρχει κίνδυνος ε, υποτροπής δεδομένου του υψηλού ποσοστού της ενεργείας και των ε, κρεμών δυσκολιών του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γι' αυτό οι Υπουργοί Οικονομικών ε, του G20 που συναντήθηκαν στο Λονδίνο στις αρχές του μήνα συμφώνησαν εν ώψη τη Συνόδου Κορυφή του Πίτσμπορκ να διατηρήσουν προ το παρόν τα, μέτρα, τα οικονομικά μέτρα στήριξη, ε, χαράζοντα μια συντονισμένη πολιτική διεξόδου από την χρηματοπιστωτική κρίση. Και οι δύο σύνοδοι κορυφή του G20, της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου, είχαν αποφασιστική σημασία για τον καθορισμό ενός συνολικού προγράμματος μεταρρύθμισης του προγράμματος οικονομικής ε, εποπτείας, χρηματοπιστωτικής εποπτείας και ρύθμισης βρισκόμαστε, βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σημείο καμπής μετά από τρεις δεκαετίες που χαρακτηρίστηκε από την απορρίθμιση και τις θεωρίες για, την για το υποτιθέμενο το χαρακτήρα των χρηματοπιστωτικών αγορών. Στην Ουάσιγκτον οι χώρες του G20 έθεσαν τα θεμέλια και καθόρισαν τις αρχές και το πρόγραμμα προκειμένου να υποβάλουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε μια πιο στενή επιτήρηση και εποπτεία και μια πιο αυστηρή ρύθμιση, ώστε να μην μένουν ζώνες προϊόντα ή χρηματοπιστωτικοί παράγοντες εκτός του πεδίου της ρύθμισης και της εποπτείας. Επίσης, οι αρχές θα πρέπει να συντονίζονται και να συνεργάζονται με στενότερο τρόπο για να αποφευθεί η αναποτελεσματικότητα μερικές φορές των εθνικών συστημάτων μια και το σύστημα είναι παγκοσμιοποιημένο και οι χρηματοπιστωτικές ε, δραστηριότητε έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Στη διάσκεψη κορυφής του Λονδίνου τον Απρίλιο ε, έγιναν πολύ σημαντικές πρόοδοι για την έμπρακτη εφαρμογή αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, λογιστικοί κανόνες ε, για τις χρηματοπιστωτικές οργανώσεις, την ανάγκη διαφάνειας ε, για τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά και τη ρύθμιση των hedge funds και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανώσεων, επίσης η ρύθμιση των αγορών χρηματοπιστωτικών παραγόντων ή η ρύθμιση των κανόνων που ισχύουν για τις ε, αμοιβέ ε, των ε, διευθυντών τραπεζών και των traders, καθώς και των πρίμα που λαμβάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε εις πέρας όχι μόνο ένα σημαντικό καθήκον προώθησης αυτών των συμφωνιών σε επίπεδο G20, αλλά ανέλαβε την αποστολή της έμπρακτης εφαρμογής αυτών των συμφωνιών, κάτι που προϋποθέτει έντονο συντονιστικό έργο το, τους τελευταίους 12 μήνες. Μερικές προτάσεις ήδη εγκρίθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο, αλλά άλλες ε, συνεχίζουν την πορεία τους στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αλλά μέχρι το τέλος του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει μια συμπληρωματική ε, δέσμη μέτρων και αποφάσεων και να προτείνει την ε, σύσταση Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου και τη σύσταση τριών ε, ευρωπαϊκών αρχών μικροεποπτείας ευρωπαϊκής κλίμακας μετά τις συστάσεις της έκθεσης Ντελαροζιέρ που ενστερνίστηκαν και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, η Αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα χρηματοπιστωτικών μεταρρυθμίσεων και μάλιστα ε, την εβδομάδα αυτή ο πρόεδρο Ομπάμα χαρακτήρισε αυτό το πρόγραμμα ω προτεραιότητα των εργασιών του. Γιατί α μην ξεχνούμε ότι στη ΣΥΠΑ ξεκίνησε αυτή η κρίση. Υπήρξε σημαντική πρόοδο ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει αυτέ. Θα πρέπει όμω. Ε, να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξει ρυθμιστική σύγκληση μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Αυτή η ρυθμιστική σύγκληση θα χρησιμεύσει και στο μέλλον ώστε να αποφευθούν σημαντικές τρευλώσεις στην αγορά. Στο Pittsburgh, εκτός ε, από την αξιολόγηση των μέχρι τώρα ρυθμίσεων και την θέση σε ισχύ των νέων μέτρων, θα πρέπει να δοθεί και ένα σαφές πολιτικό μήνυμα θα πρέπει να εκφραστεί η βούληση των κρατών, των πολιτικών ηγετών, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να χαραχθεί ένα στέρεο ρυθμιστικό πλαίσιο με αποτρεπτικό χαρακτήρα, ώστε κανείς να μην διανοηθεί από τη στιγμή που θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση ότι θα επαναληφθούν οι προηγούμενες πρακτικές που αποτέλεσαν το γενεσιουργό αίτιο της κρίσης και όλα αυτά να γίνουν σαν να μην είχε συμβεί τίποτα στο παρελθόν. Γι' αυτό θα απαιτηθούν ε, εγγυήσει και ο σεβασμός κανόνων από όλου. Ο σεβασμός των κανόνων ιδιαίτερα για τις αμοιβέ που ίσως ε, ξαναφέρουν σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πραγματική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και υποστηρίζει σύσσωμη αυτή τη δέσμευση. Και μάλιστα όλα αυτά τα θέματα βρίσκονται ε, ως προτεραιότητα σε πολλά προγράμματα και κυρίως στο θέμα της ε, μεταρρύθμισης ε, των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Στο Λονδίνο έγινε ένα τεράστιο άλμα πρόοδου για τα ιδρύματα αυτά, αλλά και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και αυξήθηκε κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ το, η πιστοτική δυνατότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οπότε το όριο είναι 750 δισεκατομμύρια δολάρια η πιστοτική δυνατότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επίσης, ε, αποφασίστηκε η κατανομή μεταξύ των διαφόρων χωρών ε, του, του Ταμείου ε, η κατανομή των δικαιωμάτων σε ύψους 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, αυξήθηκε η χρηματοπιστωτική ικανότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ώστε να μπορεί να χορηγεί περισσότερα δάνεια στις ε, φτωχότερες χώρες. Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Και το τελευταίο εξάμεινο έγινε πολύ σημαντικότερη πρόοδος από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια συμφώνησε να συμβάλλει στο μέτρο των δυνατοτήτων και των ευθυνών της στην αύξηση των ε, κονδυλίων του Ταμείου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μάλιστα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να προσθέσουν στις ε, συνηθισμένες τους ε, ε, εισφορές 125 επιπλέον δισεκατομμύρια προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η πραγματοποίηση των νέων στόχων. Οι ηγέτες των G20 θα ζητήσουν αύξηση της παρουσίασης των κυβερνητικών οργάνων στις διάφορες εποπτικές οργανώσεις. Φυσικά, οι αναδυόμενες οικονομίες διεκδικούν πιο ίση και δική εκπροσώπηση. Το υποστηρίζουμε αυτό, αλλά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες που θα υλοποιούν αυτή την ε, εκπροσώπηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί, όπως ε, πιστεύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι η καλύτερη εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στα όργανα αυτά είναι μια ενιαία εκπροσώπηση. Α μην ξεχνούμε και την προετοιμασία τη διάσκεψη κορυφή τη Κοπεχάγη για το περιβάλλον. Ε, έχουμε και την ανάγκη επανάληψη των διεθνών ε, εμπορικών συμφωνιών, χωρί να ενδώσουμε σε προστατευτικού ε, πειρασμούς, σε πειρασμού προστατευτισμού και να μην ξεχνούμε και τι πιο ευάλωτες χώρε που πολύ πιο δύσκολα θα υπερβούν την κρίση. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μία ανακοίνωση με θέμα τι κλιματικέ αλλαγέ. Τέλος θα ήθελα να σας επισημάνω την δεδηλωμένη βούληση τη, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ, του Συμβουλίου μάλλον το G20, εν της Συνόδου Κορυφής του Pittsburgh, να τεθούν τα θεμέλια για μια πιο αηφόρο οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποιες στρατηγικές διεξόδου, άμεση εφαρμογής, αλλά εφαρμογής τους την κατάλληλη στιγμή και με συντονισμένο τρόπο. Ο καθορισμός τέτοιας στρατηγικής θα είναι κεφαλαιόδου σημασία όχι για να ξεφύγουμε από την κρίση και να μείνουμε στο πυρόβλητο της κρίσης, αλλά για να υλοποιήσουμε και έναν ορίζοντα μέσο πρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αηφορίας και για τα δημόσια οικονομικά, για τα επίπεδα απασχόλησης, αλλά και για την δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Θα ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους των ε, πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέρους του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος δηλαδή, λαμβάνει το λόγο η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ Μάρτσα, κύριε Επιτροπέ, Βελμονιά βρισκόμαστε ενώπιον μια διεθνού κρίση, γιατί ο χρηματιστικό τομέα δρά διεθνώ και θα πρέπει και εμεί κατά το δυνατόν να υιοθετήσουμε διεθνώ δεσμευτικέ λύσει. Και αυτό είναι τόσο σημαντική η διάσκεψη κορυφή του G20 στο Pittsburgh η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει βέβαια και εκείνη να δράσει, θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της σε μια ισορρόπηση μεταξύ της ελευθερίας και της υπευθυνότητας. Αξίες που είναι η βάση για τη δική μας κοινωνική ε, οικονομία αγοράς και το επίκεντρο του δικού μας ε, προγραμματισμού στο ΕΛΚΑ. Το G20 είναι πολύ σημαντική διάσκεψη, ε, αφορά περισσότερο από ένα όραμα όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό. Να έχουμε περισσότερη διαφάνεια, καλύτερους κανόνες για την επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κύριε Επίτροπε ε, Αλμούνια, είπατε ότι υπάρχουν προτάσεις για τα hedge funds. Τι θέλετε να πετύχετε στον τομέα αυτό, στο J20. Μια γλίγορη μεταρρύθμιση και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αυτό πρέπει να επιτευχθεί. Το είπατε κι εσείς θα πρέπει να εργαστούμε εγκαιρά σε συντονισμένη πολιτική εξόδου και να μην δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Πρόεδρε τα συστήματα των ε, ε, δώρων των, για, τους, ε, για το ανώτατα στελέχη των τραπεζών να αλλάξει γιατί απειλείται η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων από αυτά θα πρέπει να δειχθούμε αποτελεσματικοί. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η διάσκεψη κορυφή του G20 θα μπορεί να επιτυχεί μόνο εάν υπάρχει σωστή συμφωνία. Αναφέρθηκα στα, χρηματοπιστωτικά. Το θέμα των κλιματολογικών αλογών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προετοιμασία τη διάσκεψη κορυφή του Σκοπενχάγη. Ε, καταπολέμηση του προστατευισμού προ όφελο τη απασχόληση. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Όλοι μαζί θα πρέπει να ηγηθούμε των αλλαγών αυτών. Αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει όλα τα ευρωπαϊκά μέλη να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να σεβαστείτε το χρόνο σας. Εκ μέρους της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει ο κύριος Μπούλμαν. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πιο σημαντικό είναι αυτό με το οποίο θα αρχίσω. Στη σημερινή οικονομική κατάσταση δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε όπως μέχρι τώρα. Γιατί θα έχουμε μόνο πολύ αργές, ε, αργούς ρυθμούς ανάκαμψης, δραματικά αυξανόμενη ανεργία και εδώ στην Ευρώπη και γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε τολμηροί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα του Κοινοβουλίου προς εσάς που θα πάτε στο Πίτσπορκ. Άκουσα πολλά ενδιαφέροντα στην ομιλία σας κύριε Αλμούνια. Θα ήθελα να συγχαρώ. Τώρα τολμήστε αυτά να τα μεταφέρετε στην πράξη. Θα πρέπει παντού όπου στο, στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές ο κερδοσκόπος είναι εκείνος που κερδίζει έναντι εκείνων που θέλουν να επενδύσουν μακροπρόσθεσμα για καλές θέσεις απασχόλησης, για καλά προϊόντα για επιβίωση των επιχειρήσεων. Εκεί θα πρέπει να βασιστείτε. Και είναι σωστό να πείτε όχι επικίνδυνοι ε, δράστες ή ε, χώροι ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να παραμείνουν ανεξέλεκτοι. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχουμε αμφίβολα προϊόντα αυτού του τύπου στην αγορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για όλους. Και μη φοβηθείτε τη συζήτηση και για τη φορολογική πολιτική. Δεν απαγορεύεται ένα διεθνές φόρο για την κίνηση κεφαλαίων θα, μπορούσαμε να τον επιβάλλουμε και να είναι προς όφελος όλων το θέμα του συντονισμού και της ευρωπαϊκής οικονομικής, ε, οικονομικής πολιτικής είναι σημαντικό. Να συζητήσουμε το θέμα της εξόδου, αλλά το σημαντικότερο είναι το θέμα της εισόδου σε μια καλή υποστήριξη της ε, οικονομίας και καλύτερο συντονισμό των οικονομικών μας πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους των φιλελευθέρων. Το λόγο έχει η κυρία Σίλβια Γκουλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Εκτιμούμε όλες τις προσπάθειες που αναφέρατε που ήδη προχώρησαν αρκετά μακριά, θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε μια υλοποίηση κάποιων στοιχείων και δεσμεύσεων των G20. Κυρίω επιστώ την προσοχή σα επί τη διαφορά μεταξύ των στοιχείων, των ενθαρρυντικών μάλλον, στο χρηματοστικό τομέα και των φρικτών στοιχείων για την ενεργεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχουμε βιώσιμα διαρκώς ανεργία θα έχουμε ανθρώπινο δράμα καταρχάς και προβλήματα στα δημοσιονομικά και έλλειψη ανάκαμψη τη κατανάλωση. Εμεί ελευθέρωσαμε ένα σενάριο αλλά ιαπωνικά μικρή ανάπτυξη, πιο ήπια ανάπτυξη σε ψηρά ετών. Βοηθήστε μα λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την εμπειρία σα, κύριε Υπουργέ, από τη Σουηδία. Έχουμε τρία πράγματα που εξετάσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διεθνή συνεργασία καταρχά. Θα πρέπει να συνεχιστεί η καταπολέμηση του προστατευτισμού. Θα πρέπει να ενισχύσουμε του διάφορου παγκόσμιου θεσμού, όπω το Παγκόσμιο Ισμικό Ταμείο. Δεν θα τα καταφέρουμε μόνοι μα και θα πρέπει συνεχώ να το στέλνει αυτό το μήνυμα η Ευρώπη. Θα πρέπει δεύτερον να υπάρχει σωστή αποτελεσματική εποπτεία και εξυγίανση τραπεζική πολύ πιο ε, λεπτομερή και α είμαστε καχύποπτοι για τι ε, ένα των ανακοινώσεων των G20. Υπάρχει το εκτελεστικό, αλλά υπάρχει και νομοθετική δουλειά πρέπει να γίνει. Και για εμά, κύριε Αλμούνια, οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εποπτεία είναι ένα βήμα προ σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Μακροπρόθεσμα θέλουμε πιο ευρωπαϊκά μέτρα θα πρέπει να σκεφτούμε κοινέ στρατηγικέ για τη διέξοδο από την κρίση, διατηρώντα το προστατεύοντα το ευρώ, να μην ε, η κοινή νομισμα... νομισματική πειθαρχία να μην υποφέρει ο κύριος Αλμούνια καλά είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στα διεθνή βήματα συζητήσεων. Θα πρέπει να προσθέτουμε την κοινοτική μέθοδο. Βασιζόμαστε πάνω σα να φροντίσετε να μην υπάρχουν μόνο οι μεγάλε χώρε που κάνουν ακουστή τη φωνή του, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακούγεται και να γίνεται εισακουστή στην παγκόσμια οικονομική αγορά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερω γιατί τηρήσατε και το χρόνο σα. Εκ μέρους των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριος Σβέν Γκίγκολτ. Ε, Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για την ομιλία σας. Έχω αρκετές ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα, η Επιτροπή Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου συνέταξε πρόταση ψηφίσματος και παραθέτω. Σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η κρίση που έχει κοστίσει πολλά σε ανθρώπινο επίπεδο και έχει καταστρεφικέ συνέπειε στου ευάλωτου στι φτωχότερε χώρε και αναμένεται αύξηση κατά 23 εκατομμύρια ανέργου. Και πάνω από 90 ε, εκατομμύρια πολύ φτωχού θα έχουμε μέχρι το 2009. Και 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν πληγεί από το AIDS και 200.000 με 400.000 περισσότεροι θάνατοι παιδιών κατά μέσο όρο στο διάστημα 2009-2015. Δυστυχώς αυτή η πρόταση ψηφίσματος δεν πέρασε παρόλο που συνετάχθη από όλες τις ομάδες του Κοινοβουλίου και το καταγγέλουμε αυτό, θεωρούμε ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το σώμα να μην μπορέσει να συντάξει ένα ψήφισμα για τους G20 όσον αφορά τα αναπτυξιακά θέματα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς να χρηματοδοτηθούν οι συνέπειες της κρίσης. Και εκεί ο Γερμανός Υπουργό Οικονομικών μαζί με την Καγκελάριο πρότειναν στο G20 να συζητηθεί η πιθανότητα ενός διεθνούς φόρου συναλλαγών Ρωτώ να μου πει η, Υπουργός και η Προεδρία του ε, Συμβουλίου υποστηρίζεται αυτή την πρόταση. Τι λέτε κύριε Επίτροπε. Δεύτερον, η φορολογική παράδοση. Οι G20 θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κατά περίπτωση μέσω ανταλλαγή πληροφοριών. Ξέρουμε ότι αυτό δεν πάει λειτουργήσει. Η Επιτροπή Ανάπτυξη πρότεινε μια καταχώρα, ένα καθεστώ αναφορά κατά χώρα, ώστε οι διεθνεί επιχειρήσει θα πρέπει να στέλνουν εκθέσει και αναφορέ κατά χώρα και προτείνουμε να εισαχθεί αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ούτω ώστε να υπάρχει πραγματική ροή πληροφοριών μεταξύ χωρών. Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα χρειάζεται διαφάνεια. Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση σα επί των συγκεκριμένων προτάσεων για να βγούμε από την κρίση και για τη χρηματοδότηση των συνεπειών τη κρίση. Σα ευχαριστώ και σα θέλω παρακαλώ χρόνου φίδου. Μην ξεπερνάτε το χρόνο, το χρόνο σας. Εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών το λόγο κύριο η κυρία Σουίνμπερν, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για τι ομιλίε που ακούσαμε σήμερα και ευχαριστώ άκουσα και την ομιλία τη κυρία Μάλστρομ για την σύνοδο κορυφή του Πίτσμπουργκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν κάποια μέτρα και κάποια οικονομισμοί στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή οι χώρε δαπανούν τεράστια ποσά για να δώσουν ενάγματα στην οικογέ... στις οικονομίες τους. Οι δύο πιο πολύπλοκες δομές του κόσμου, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να αναθεωρήσουν όλη τους την, την δομή της οικονομίας. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έξοδος από την από την κρίση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο διακανονισμού για να μην δημιουργηθούν δυνατότητες για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για κάποιες μεμονωμένες χώρες. Δεν θα υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα. Συνονισμό, συνοσμένη προσέγγιση είναι η μόνη δυνατότητα για να βρούμε τους πόρους που χρειάζονται σε όλη την Ένωση εάν οι τράπεζες που, χρειαζ... που στις οποίες βασόμαστε χρειάζονται τόσο κεφάλαια που οι φορολογούμενοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβουν πολύ περισσότερο κοινού, δεν θα μα ευχαριστήσει κανένα για όλε αυτέ τι εξελίξει. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί διεθνή συντονισμένη προσέγγιση και να διατηρηθεί για να εξασφαλίσουμε μελλοντική πρόσβαση σε κεφάλαιο παντού στην Ουαλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τις παρεμβάσεις που θα διαρκέσουν μόνο ένα λεπτό εκ μέρους της Γκούε, Το λόγο έχει ο κύριος Μιγγέλ Πόρτες. Ευχαριστώ. Στην Πορτογαλία τα κέρδη των τραπεζών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν κατά 18%. Ακόμη περισσότερο, μόνο η ανεργία ξεπέρασε αυτό το ποσοστό. Και μάλιστα η Πορτογαλία αυτή τη στιγμή είναι υπόδειγμα αποτυχημένης υπόσχεσης που έγινε από το G20 και ήταν μια απόπειρα ε, διεξόδου από την κρίση με μια νέα οικονομική παγκόσμια τάξη. Λάθος. Ανακριβές. 50 εκατομμύρια νέων ανέργων και 200 εκατομμύρια νέων νεόπτωχων ε, είναι απόδειξη της ε, εσφαλμένης αυτής και θετημένης υπόσχεσης. Η κυρία Υπουργό μα είπε ότι ασχολούνται με τα πριμ και τα hedge funds. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο θα πρέπει να μιλήσουμε για το τέλος των φορολογικών παραδείσων, για, για τα ποσοστά επί των διασυνοριακών συναλλαγών. Θα πρέπει να μιλήσουν για το τέλος του τραπεζικού απορρίτου. Αυτά θέλουν να ακούσουν οι άνθρωποι, ο κόσμος. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Ευρώπης ε, Ελευθερίας και Δημοκρατίας, ο κ. Μποργέζιο. Ευχαριστώ. Οι λαοί τι πίστη μπορούν να έχουν σε μια ρύθμιση των χρηματοδοτικών αγορών που ανατίθεται στους ιερείς των παγκόσμιων ε, οικονομικών ναών. Στην Αμερική έγινε μια λαϊκή εξέγερση, μια νέα επανάσταση συντηρητική των λαών κατά της οικονομικής ολιγαρχίας. Εμείς οι λαοί δεν πιστεύουμε στις πολιτικές διάσωσεις των οικονομικών ισχύων που κάνουν το φορολογούμενο να πληρώνει στην Αμερική όπως στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα έπρεπε να δώσουν πόρου στην πραγματική οικονομία, να ασχοληθούν με την παραγωγή, με την εργασία. Τα αποτελέσματα των G20 τι βλέπουμε πέρα από τον πόνους και την εξάλληψη των φορολογικών παραδείσων. Οι παρεμβάσεις έχουν σαν σκοπό να προστατεύσουν αυτούς που δημιούργησαν αυτή τη φούσκα την οικονομική. Πολλά χρήματα δίνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χρήματα από την οικονομία μα που δίνονται στου υπεύθυνου των ε, φυσαλίδων αυτών των οικονομικών. Δο, μόνο 50 δισεκατομμύρια δόθηκαν από τα πολλά χρήματα που δόθηκαν, διαθέθηκαν για την απάλυνση των οικονομικών συνεπειών. Και στη ΣΥΠΑ και στην ε, Ευρώπη σαν σερβιτόροι των οικονομικών δυνάμεων κινούνται οι πολιτικοί. Ξύπνα Ευρώπη. Ακολούθα το παράδειγμα του Αμερικανικού λαού που ξεκινά μια δεύτερη μεγάλη επανάσταση, την επανάσταση συντηρητική του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Να σας υπενθυμίσω ότι καλό θα ήταν να τηρήσουμε το χρόνο αγόρευσης που είναι ένα λεπτό. Διαφορετικά θα αναστατωθεί το πρόγραμμά μας αν δεν τηρείτε το χρονοδιάγραμμα. 1,5 λεπτό ο Hans Peter Martin. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε χρειαζόμαστε μια επανάσταση της δημοκρατίας. Αυτό διαφαίνεται ιδιαίτερα σε αυτή τη διαδικασία που ευτυχώς τώρα κινήθηκε. Ε, και οι J20 μπορεί να γίνουν και παραπάνω, θα μπορούσε να φανταστεί κανένα και έναν άλλο αριθμό. Πώς σκέφτεται η Κομισιόν να προωθήσει ένα δημοκρατικό μηχανισμό ελέγχου. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο, αλλά αυτό που προωθείται χρειάζεται ένα δημοκρατικό έλεγχο από εκλεγμένου βουλευτέ σε μεγαλύτερο πλαίσιο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα επίση να αναφερθώ ρητά στο θέμα του συστημικού προβλήματος που θα πρέπει να εξεταστεί, δηλαδή το θέμα των προβλημάτων που ξεκίνησε με την Λέιμαν, με τα προβλήματα των ε, υποθηκών κλπ. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ότι ορισμένες δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν γίνει πολύ μεγάλες για να τους επιτρέψουν να αποτύχουν. Όσον αφορά το θέμα του τι είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο του 99 την ομάδα του φόρου Τόρπιν χρειάζεται οπωσδήποτε να δράσουμε ευρωπαϊκά, να μην αφήσουμε να μας πιέσουν εκείνοι που δεν θέλουν τη σωστή Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε τους υπόλοιπους αγορητές. Πρώτος ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία βελτιώνονται. Οι πολλοί λόγοι της κρίσης δεν έχουν εξαλειφθεί όμως ακόμα τελείως και γι' αυτό η πολιτική βούληση δεν θα πρέπει να μειωθεί ούτε η αποτελεσματικότητα και η τόλμη των αντίων. Σήμερα συζητάμε για το G20. Καλή διαδικασία αυτή. Χρειάζομαστε νέες καλύτερες δομές ελέγχου των προτεραιότητων ε, χρηματοπιστωτικούς ε, ελέγχους για την ε, επίτευξη της κοινωνικής ε, δικαιοσύνης στον κόσμο. Υπό τρεις Η δημιουργία της κοινοβουλευτικής διαδικασίας επικύρωσης περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη στον κόσμο, δηλαδή τα εξαγόμενα προϊόντα μας είναι οι, αρχές, οι αρχές και αξίες ε, των, ε, της χάρτας βασικών δικαιωμάτων και τρίτον θα ήθελα σε εκείνους τους τομείς στους οποίους η J20 δεν μπορεί να πετύχει συνένεση να έχουμε ευρωπαϊκούς δεκανοσμούς που χρειάζονται. Λέμε ναι σε μια ευρωπαϊκή επιτήρηση των χρηματοπιστωτικών αγορών λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η έκθεση Λαροζιέ είναι λίγη, λέμε ναι στη συζήτηση για τα, τις πληρωμές των πόνους αυτών, εμείς θα πρέπει να ε, τροποποιήσουμε την βάση υπολογισμού και όπου υπάρχει ένα πόνους θα πρέπει να υπάρχει και ένα μάλλον, ένα μείον, να μπορούν να προωθούν για τα έτη 2009 και 2010 να μειώσουμε τα κύρια στοιχεία της κρίσης, δεν θα πρέπει να μειωθεί η πολιτική βούληση και μετά την ομιλία σας περνάμε με αισιοδοξία στο Πίτσπορκ. Κύριε Περβάνος Μπέρες, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία εκπρόσωπε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, ένα χρόνο μετά την πτώχευση τη Lehman Brothers, η φωνή που θα εκφράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Pittsburgh ε, θα είναι κρίσιμη. Αν δεν θέλουμε να ξαναρχίσει η κρίση και να παραμείνει ε, αδιάλειπτη η ορμή της βελτίωσης. Πέρσι τον Απρίλιο τη Σύνοδο Κορυφή του G20, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύθηκαν να αυξήσουν τα μέσα ε, και τα κονδύλια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Υπήρξε κινητοποίηση για την υλοποίηση αυτού του στόχου, αλλά πολύ φοβούμε ότι αυτή η προθυμία ε, κρύβει την ε, απροθυμία να προωθηθεί η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επίσης θα πρέπει να γίνουμε θύματα της μόδας, γιατί ακούμε παντού για τα αστρονομικά πριμ των διευθυντών και των traders ε, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ένα σύστημα που θα ε, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη επένδυση. Αλλά αυτό θα πρέπει να αποσπά την προσοχή μας από το μείζον θέμα των φορολογικών παραδείσων, κυρίως θέμα της ε, διάσκεψης του Λονδίνου. Όπως είπε και ο κύριος Μπούλμαν, Βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πώς οι τράπεζες θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της διεξόδου από την κρίση για να γίνει η επανάληψη της συζήτησης ε, για τη φορολόγηση των συναλλαγών. Γιατί και από εκεί θα μπορούσαμε να εκμεύσουμε κάποια κονδύλια για να ενισχύσουμε τις μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις. Γιατί στηρίχθηκαν οι τράπεζες από τα κράτη για να ξεφύγουν από την κρίση. Είναι δίκαιο λοιπόν και λογικό και αυτές τώρα να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση και την αναζωογόνηση της οικονομίας. Επίσης όταν εξετάζουμε το θέμα της ανεργίας, από την αρχή τους, οι σύνοδοι κορυφή του G20 είχαν μια δυναμία και ένα κενό, γιατί ασχολή, δεν ασχολήθηκαν με το συνολικό αντίκτυπο προς την ανεργία και την επαναφορά μιας στρατηγικής που θα επιτρέψει τη διόρθωση των ανισορροπιών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βολφ Κλίντς. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζω την γρήγορη και αποφασιστική αντίδραση της ομάδας των G20 ε, φαίνεται ότι έχουμε σβήσει τη φωτιά, αλλά τα θεμέλια δεν είναι ακόμα σταθερά γιατί ε, οι προείδες έχουν εντύπωση ότι κοινωνικοποιούνται τα, οι απώλειες. Κοιτάξτε, ακούμε πολλέ ομιλίε, αλλά δεν κάνετε αυτό που θα πρέπει να κάνετε, να υποστηρίξετε λίγο την πραγματική οικονομία. Η ιδεολογία και η ευθύνη είναι κάτι που έχουν εξαφανιστεί, νομίζω. Ελπίζω οι, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουν ενωμένα. Χρειάζονται νέε δομέ, ε, καλύτερα ε, ίδια κεφάλαια, κίνητρα, μακροπρόθεσμα, όχι βραχυπρόθεσμα, συντονισμένη στρατηγική, περιορισμό του προστατευτισμού και μείωση του και λύση του προβλήματος too big to fail. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κορνέλης Δεγιόγκ είναι ο επόμενος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέχρι τώρα οι G20 επικεντρώθηκαν σε μέτρα για τον χρηματοστατικό τομέα. Όμω όλοι φαίνεται να ξεχνάνε ότι επίση και η πραγματική οικονομία υποφέρει από την απληστία και την επιθυμία βραχυπρόθεσμων κερδών. Έχω κάθε σεβασμό για τι μικρέ επιχειρήσει παρά τι αντικσότητε που θέλουν να επιβιώσουν. αξίζει να πάρουν τα δάνεια που δικαιούνται. Όμω δεν έχω κανένα σεβασμό για τη διοίκηση μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δεν έχουν καμία επαφή με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν και μόνο σκέφτονται την ανάπτυξη, την κερδοσκοπία. Γι' αυτό ζητώ από τους g να συζητήσουν τρόπους να γίνει πιο δημοκρατική οικονομία να εξασφαλίσουμε ότι εντό τη επιχειρήσεω οι εργαζόμενοι και άλλοι που εκπροσωπούν τα γενικά συμφέροντα έχουν αρκετή εξουσία για να ελέγχουν τη διοίκηση. Εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το καθεστώ για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση, το καταστατικό αυτή. Θα πρέπει να είναι αδύνατον η μέτοχη και η διαχείριση να αναπτύσσονται μέσω κερδοσκοπία ει βάρο των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των επιχειρήσεων και εκείνων που εργάζονται εκεί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κριστίνα Μορβάη, η επόμενη μιλήτρια. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν είναι τραπεζίτες και επικεφαλής επιχειρήσεων. Μικροί γεωργοί, μικροί επιχειρηματίες, ε, δημόσιοι υπάλληλοι είναι. Η, η Ευρώπη έχει βαρεθεί, η πλειοψηφία της έχει βαρεθεί με το παρόν σύστημα. Όπου οι πολυεθνικές και οι τράπεζες κυβερνούν τον κόσμο χρειάζονται και θέλουν ένα νέο παράδειγμα που πρέπει να δημιουργηθεί. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή από παγκοσμιοποίηση προς τοπική διοίκηση και παραγωγή. Οι αποφάσεις τα λαμβάνονται μην λαμβάνονται βάση του κέρδους, αλλά βάση των αποφάσεων ένα άνθρωπος. Να ξεφύγουμε από τον ΠΟΕ και τη γεωργία, να φτάσουμε στην ασφάλεια τροφίμων και τοπική παραγωγή τοπική καλλιέργεια. Παρακαλούμε στο G20 να εκφράσετε την άποψη της πλειοψηφίας της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά το λόγο έχει ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποιος θα πρέπει να διακανονίζει ποιον και πώς. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα στην διάσκεψη κορυφή του G20 και αν υπάρχει συμφωνία ότι δεν θα πρέπει να ξαναπεράσουμε σε αχαλήνεωτες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό κομμάτι, ο τρόπος του διακανονισμού είναι ακριβώς ακόμα ανοιχτών. Ε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε για το ίδιο κεφάλαιο για τους ε, επιχειρήσεις rating τι θα γίνει επίσης με κάποια προϊόντα και την έγκρισή τους αλλά και το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού για, τα, για το φόρο, για τον έλεγχο θα υπάρχει ε, επίσης ε, διαφωνία όσον αφορά τα μπόνους αυτά και όσον αφορά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγει ένα φόρο Τόρμπιν. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ καλά προτυπωσμένοι όταν πηγαίνοντας στο J20 και νομίζω ότι η Κομισιόν τη ζωστή άγουσα που δεν ε, εξαρτάει αυτόν από το τι θα κάνουν οι άλλοι. Δεν θα πρέπει κανένας δράση, κανένα προϊόν, καμία θέση χρηματοπιστωτική ε, να είναι χωρίς έλεγχο. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα της γενικής ανάκαμψης της οικονομικής και δεν επιτρέπεται να συνεχίσουμε όπως το παρελθόν προωθώντας τις <clears throat> ανισορροπίες στον κόσμο υπέρ της, των ΙΠΑ και των μεγάλων βιομηχανικών χωρών. Θα πρέπει να δούμε πώς θα επιλύσουμε τα προβλήματα της φτώχειας και της πείνας στον κόσμο και από εκεί ελπίζουμε για αυτά τα θέματα να υπάρχουν ε, ενάσματα από την J20. Κάτι δεν τα έχει συζητήσει αυτά τα θέματα εκτός από τον κύριο Αλμούνια. Θα πρέπει να τηρήσουμε την Συμφωνία Σταθερότητας και Ανάπτυξης στην Ευρώπη. Επειδή την έχουμε, την έχουμε αναθεωρήσει τη συμφωνία αυτή, γι' αυτό καταφέρουμε να είμαστε ε, σε θέση να δράσουμε στην Ευρώπη. Και αυτό θα επιτρέψει μια γλίγορη στρατηγική εξόδου από τα υπερβολικά χρέη και σε μια πολιτική ανάκαμψη πραγματική. Ευχαριστώ. Τώρα κύριος Έντουαρτ Σίκλον. Ευχαριστώ Πρόεδρε διαβάσαμε στον τύπο ότι το κυρίως θέμα του G20 θα είναι τα πριμ των ναι. διευθυντών τραπεζών. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Γιατί άρρυψη και δινεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι λογικό να υπάρχει εποπτεία αργότερα και έλεγχος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τεράστιες ανισορροπίες στο εξωτερικό εμπόριο και αυτές οι ανισορροπίες αποτέλεσαν το αίτιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε συνδυασμό με κάποιες εσωτερικές επίσης ανισορροπίες. Επίσης θα πρέπει να ελέγξουμε ε, την εφαρμογή των μέχρι τώρα αποφάσεων και αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Θα χρειαστεί να περάσει και μια διετία για να δούμε ποιες ήταν οι αλλαγές στο ΑΕΠ από τα νέα μέτρα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς εφαρμόστηκαν τα πακέτα με τα ενάψματα. Κατάφεραν να αναζωογονήσουν την οικονομία. Πρέπει να περιμένουμε λίγο χρόνο για να διαπιστώσουμε αν υπήρξαν όντως θετικές αλλαγές. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι συνεπής και να εξακολουθεί να επιμένει στη μείωση του δημοσιονομικού έλλειμματος. Παρακαλώ να μην ξεπερνάτε το χρόνο σας γιατί είναι περιορισμένος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι ο επόμενος ομιλητής. Ένα λεπτό. Με κεντρικό θέμα τη διαχείριση των πόνους δεν ακουμπά σε καμιά περίπτωση τη ρίζα του προβλήματος και δυστυχώ δεν αποτελεί βήμα προς τη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος. Η σειρά προτάσεων για τροποποίηση των κανονισμών περιορίζεται στην ανάλυση επιφανειακών ζητημάτων και δεν επικεντρώνεται στους κοινωνικούς στόχους. στόχος θα έπρεπε να είναι η συνολική χρηματοπιστωτική αλλαγή ο δημόσιος και κοινωνικός έλεγχος μια πιο δημοκρατική σύνοδος που θα ενέπλεκε το σύνολο των κρατών θα αντιμετώπιζε ζητήματα όπως η αυξανόμενη ανεργία οι καλπάζουσες τιμές σε βασικά αγαθά και καύσιμα θα έπαιρνε ουσιαστικές αποφάσεις για παρέμβαση στην αγορά με στόχο τον τερματισμό της συνεχούς ιδιωτικοποίησης και της καταστροφής του κοινωνικού κράτους. αυτές είναι οι πραγματικές ανάγκες των λαών. οι πολίτες σήμερα κύριε πρόεδρε απαιτούν συνολικές δομικές αλλαγές μακριά από το νεοφιλελεύθερο σύστημα που οδηγεί στην υπανάπτυξη αντί στην ανάπτυξη μακριά από τη μεγιστοποίηση της κερδοσκοπία, η οποία στρέφεται εις βάρος των συμφερόντων των λαών. Ο κύριος Γκοζές για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι για την αποφασιστικότητα που δείχνετε. Η Ευρώπη φαίνεται ότι αρχίζει και εφαρμόζει μία αποτελεσματική ρυθμίση, αλλά δεν μπορεί να μείνει απομονωμένη. Χρειαζόμαστε διεθνή συνεργασία και συντονισμό. Αυτό περιμένουμε από το G20. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εφαρμογή των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων. Γιατί το πλαίσιο ε, το διεθνές πλαίσιο θα πρέπει να ταχθεί στην υπηρεσία των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ας μην ξεχνούμε ότι η κρίση δεν ε, πέρασε, δεν θα πρέπει να επανέλθουμε στην επόμενη κατάσταση και να αποφύγουμε, θα πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε την επανάληψη της κρίσης που παραβλάβει την οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Θα πρέπει να ενισχυθεί η εποπτεία και η ρύθμιση. Είναι απαραίτητα αυτά και η ρύθμιση θα πρέπει να είναι αντάξια του συστημικού κινδύνου που επιβάλλουν οι χρηματοπιστωτικές ε, ε, οργανώσεις. Επίσης, ε, θα πρέπει να αυξήσουμε τις απαιτήσεις για τους ίδιους πόρους και να εφαρμόσουμε και διεθνώς τους κανόνες της Βασιλείας. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβέ στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, θα πρέπει η Επιτροπή Αμοιβών να επαναφέρει μια διαφάνεια αυτών των αμοιβών με πιο αυστηρέ δημοσιεύσεις και να αποφύγει τα αστρονομικά πριμ. Και η ρυθμίση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς είναι απαραίτητη. Το ίδιο και η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης και της εκπροσώπησης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτές είναι μερικές από τις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών από την επόμενη διάσκεψη κορυφής του G20. Και εκεί η Ευρώπη θα πρέπει να αποφανθεί με ενία φωνή, με ισχύ και αποφασιστικότητα. Ο Αλεχάνδρο Σέρκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πίτροπέλ Μουνιά, κυρία Υπουργέ, σας θέρμα παρακαλώ. Στο Πίτσμπουργκ δεν θα πρέπει να ξεχανάτε ότι δεν έχουμε μόνο μια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση άνευ προηγουμένου, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και μια βαθύτατη κοινωνική κρίση με ολέθριες συνέπειες ε, για τους πιο αναξιοπαθείς για ανθρώπους που έχουν μόνο μία δουλειά ή είναι μικροεπαγγελματίες ή μένουν σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές. Σημαντική είναι η οικονομία, αυτό θα πρέπει να πει το Pittsburgh, αλλά ακόμη πιο σημαντικά είναι τα άτομα και η οικονομία θα πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Επίση, το Pittsburgh δεν θα πρέπει να ξεχάσει ότι υπάρχει και Ευρώπη, θα πρέπει να ε, υψώσει τη φωνή τη γιατί έχω την ε, ε, επιστολή των τριών ε, πρωθυπουργών με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν αναφέρεται τίποτα για την Ευρώπη. Γιατί θα πρέπει να μιλήσει ενωμένη με ενιαία φωνή η Ευρώπη. Γιατί δεν αναφέρεται ούτε μία λέξη για την Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να, να ακούσουμε ξεχωριστέ φωνέ. Θα πρέπει με ενωμένη φωνή να μεταρρυθμίσουμε την αγορά και να αποτρέψουμε την επανάληψη της κρίσης στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαρθία Μαργκάγιο για δύο λεπτά. Κυρίε και κύριοι, συμφωνώ με πολλές προτάσεις των προελισσάντων. Συμφωνώ ότι είναι πολύ νωρίς ε, για να ε, αφαιρέσουμε τα δεκανίκια από τον άρρωστο, αλλά θα πρέπει να τον προετοιμάσουμε για να μπορεί να περπατήσει χωρίς αυτά. Να, να απορροφήσουμε την υπερβολική ρευστότητα των αγορών, να διορθώσουμε τις ανισορροπίες των δημοσίων οικονομικών και να βελτιώσουμε την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Πολλά θα πρέπει να γίνουν στο Πίτσμπουργκ και μόνοι μα δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε κάποιου μηχανισμού έγκαιρη προειδοποίηση. Λειτουργικού όμω, γιατί οι προηγούμενοι δεν ήταν λειτουργικοί και αποτελεσματικοί. Θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο, γιατί ούτε και αυτό λειτουργήσε σωστά. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να ρυθμίσουμε και τα πριμ και του φορολογικού παραδείσου. Όλα αυτά τα μέτρα είναι απαραίτητα, αλλά δεν αρκούν από μόνα του. Ακόμη πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, είναι να γίνουν πιο εύρωστες οι χρηματοπιστωτικές οργανώσεις, να περιοριστεί η χρέωση και να προβλεφθούν κάποια ταμεία στον καιρό των απαχιών αγελάδων για να είναι πιο εύκολη κατάσταση στην περίοδο των ισχνών αγελάδων. Ε, χαίρομαι που στηρίζεται στην έκθεση Λαροζιέρ, αλλά είναι ανεπαρκής κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα μια πιο κεντρική εποπτεία. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς συντονισμό με τα εποπτικά όργανα και των άλλων ε, σημαντικών περιοχών του κόσμου. Επίσης, θα πρέπει να γίνει κάτι και για το εμπόριο. Φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αναφιόμενες οικονομίες, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να άρουμε τους φραγμούς ε, που παρακολύουν ακόμη την, ε, το εμπόριο. Επίσης, θα πρέπει να θέσουμε τις βάσεις μιας αηφόρου ανάπτυξης και για τις επερχόμενες γενιές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανοιχτές αγορές ελεύθερες που θα ενισχύουν την καινοτομία, αλλά δεν θα είναι τελείως αρρύθμισης και ξέφραγο αμπέλι. Θα ήθελα να σας δώσω ένα στοιχείο που είναι γνωστό για τον Αλμόνια, μια παράθεση από τον Δον Κιχώτη, γιατί καλά τα λόγια, αλλά θα πρέπει να τηρούνται κιόλα. Ο Πίτερ Σκίνερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Συμφωνώ απόλυτα για αυτά που είπατε για βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να τονιστεί στους G20. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το κεφάλαιό μας για να εστιαστούμε στα πριμ των τραπεζιτών. Δεν είναι σωστό αυτό. Ούτε και ευχολόγια τη λύση των παγκοσμίων προβλημάτων μπορεί να επικρατήσει συζητήσει. Ο τομέα των χρηματοστικών υπηρεσιών καίγεται. Καταρχά, θα πρέπει να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά και θα πρέπει να παραμείνει σβηστή. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σωστή συνεπή προσέγγιση. Είναι καλό βήμα η G20, αλλά χρειάζεται και μόνιμε δομέ. Όπω το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο, να ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως τα FRS. Αν το συστημικό κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν θα πρέπει να κοιτάμε στον καθρέφτη προς τα πίσω, στο αυτοκίνητό μας, αλλά να εστιαζόμαστε στον δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πίτερ. Ο κύριο Καντέ Αρίφ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η οικονομική κρίση που περνάμε είναι διαρκεία και βαθιά και χρειάζεται, είναι απαραίτητο να γίνουν οι αναγκαίε ρυθμίσει και να υπάρχει πλαισίωση του χρηματοδοτικού συστήματο των τραπεζών και να αποφύγουμε η σημερινή κρίση να εμφανιστεί εκ νέου στο μέλλον πιο βία. Το σύστημα το οικονομικό θα πρέπει να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία και να μην συνεχίσει να την καταστρέφεται. Την άποψη, η τελευταία σύνοδο των G20 στο Λονδίνο που αναφέρθηκε, έκλεισε με προτάσει ε, μερικέ και ε, λόγια που δεν μετετράψαν σε πράξεις. Και έναντι αυτής της καταστάσεως για το Pittsburgh, για να είναι χρήσιμη η σύνοδος G20 στο Pittsburgh, θα πρέπει τελικά να επιμείνει για σωστή ρύθμιση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενωθοποιηθούν. Διάφοροι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε διάφορα στοιχεία. Θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στο θέμα της, του εμπορίου και τη ανάπτυξη. Στο Πίτσμπουργκ θα τεθεί θέμα τη ανάκαψης του κύκλου συζητήσεων τη Ντόχα να ξαναξεκινήσει υπό τον όρο που ο στόχο να είναι στο επίκεντρο του κύκλου, δηλαδή η ανάπτυξη. Και να μην μείνει παράμερα. Οι εταίροι μα του Νότου δεν θα δεχθούν σωστά ε, οι ανησυχίε του να μην βρίσκουν ανταπάντηση. Θα πρέπει τελικά να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και να τεθούν και σωστέ βάσει για τη σωστή παγκόσμια οικονομική διαχείριση στου G20. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Επόμενο αγορητή, εκείνο Χάρκ Ατόντο, που έχει το λόγο για ένα λεπτό. Κύριε, κυρία Υπουργέ, κύριε Αλμούνια, Τρεις ιδέες θα εκφράσω σε ένα λεπτό. Καταρχάς περισσότερη Ευρώπη, διότι σε, αυτό, σε αυτή την κατάσταση, την παγκόσμια κρίση, θα πρέπει να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Διαφορετικά η Ευρώπη δεν θα διαδραματίσει κανένα ρόλο, δεν θα έχει πυγμή. Και πέρα από τη δημιουργία νέας διακυβέρνησης για τον κόσμο, πέρα από το νέο ρυθμιστικό σύστημα, το νέο εποπτικό σύστημα και διεθνή, το διεθνή συντονισμό θα πρέπει να σταματήσουν η φορολογική παράδειση, να καταργηθούν. Θέλουμε να υπάρχει μια διεθνής φορολόγηση. Διεθνής φορολόγηση είναι πιο σημαντικό. Και η αγορά πρέπει να πίσω το υπόψη. Πρέπει να δούμε ποιες, ποια θα πρέπει να είναι η δεοντολογία για το εμπόριο. Χρειάζεται νέα νοοτροπία ε, εταιρική ευθύνη για, τους, για τις επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμη σημασία. Θα πρέπει η επιχείρηση να είναι ένα κομμάτι της κοινωνία. Η επιχείρηση και η εταιρεία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη έναντι των μετόχων και έναντι της ε, κοινωνία. Ευχαριστώ. Και τώρα έχουμε τη διαδικασία Catch the Eye. Πρώτη η κυρία Ντάτη. Και παρακαλώ ένα λεπτό έχετε το λόγο. τηρήσετε το χρόνο σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Υπουργέ, κύριε Αλμούνια. Στις 3 Σεπτεμβρίου η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία συμφώνησαν να, να μιλήσουμε μία φωνή και με ευρωπαϊκή συνένεση για τα θέματα της αντιμετώπισης ε, των πριμ, των traders. Το Συμβούλιο μας είπε ότι θα συνεδριάσει στις 27 για να προετοιμάσει το G20. Σας ε, παροτρύνω λοιπόν να βρείτε μία λύση για κοινή απάντηση που θα είναι φιλόδοξη για να ρυθμιστούν τα πριμ των traders γιατί στα τελευταία διάσκεψη του Απριλίου δεν τηρήθηκαν, γιατί ε, οι τράπεζες ε, έδωσαν τα κονδύλια για να ε, πληρωθούν οι αμοιβέ των ΠΡΙΜ, παρόλο που οι τράπεζες στηρίχθηκαν με κρατικές ενισχύσεις. Δεν θα καταλάβει ο κόσμος αν δεν ληφθούν κάποιες αποφάσεις στο G20. Θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν οι αδυναμίες και όταν δίνονται κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να διορθώνονται τα κενά θα πρέπει να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα και κοινά μέτρα στο Pittsburgh, διότι μόνοι μας δεν μπορούμε να είμαστε ενάρετοι. Θέλουμε καλύτερη πλαίσια και καλύτερη διακυβέρνηση και υπευθυνότητα. Επίσης θα πρέπει οι κυρώσεις να εφαρμόζονται οπωσδήποτε αν υπάρχουν παραβιάσεις ή παραλήψεις. Το λόγο έχει η κυρία Μόνικα Μπέναβα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Μάστρομ, κύριε Επίτροπε, νομίζω ότι το πρόγραμμα που προσφέρετε ήταν αρκετά φιλόδοξο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε στην ε, διάσκεψη κορυφή του g να το παρουσιάσουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα συμπεράσματα. Ε, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και να μπορεί να παρουσιαστεί και στους πολίτες. Γιατί όπως είδαμε, ακόμα το πρόβλημα δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό αναφερόμαστε στο θέμα του ελέγχου, στο θέμα της διαφάνειας που θα πρέπει να εισαχθεί. Αλλά έχω την εντύπωση ότι προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε κάποιους ε, τομείς. Δεν αναφέρεται όμως τίποτα για τον έλεγχο των manager. Δεν αναφέρεται τίποτα ότι δεν θα ξεκινήσει ο μηχανισμός αυτός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυξάνεται η ανεργία, ότι έχουμε προβλήματα στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να περιοριστούμε στα θέματα που μπορούμε πραγματικά να εφαρμόσουμε στην πράξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα Κάμφιν, ένα λεπτό. Bonjour. Vous, vous avez parlé... Χαίρετε. Αναφερθήκατε στη διοίκηση του Διεθνούς Νομισματικού Τομείου δεν ξέρω, στους, ε, στην ομάδα των 20 θα αναφερθεί στο θέμα των όρων που επιβάλλονται από το Διεθνές Νομισματικό Τομείο στους ε, χώρες ε, όταν τους δανείζουν χρήματα. Γιατί είδαμε ποιες είναι οι επιπτώσεις σε κάποιες χώρες. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό και ποια είναι η θέση της Κομισιόν και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινέζικη πρόταση να υπάρχει ένα διεθνές νόμισμα που να είναι κάπως διαφορετικό για να ελέγχεται καλύτερα το διεθνές ε, νομισματικό σύστημα αντί του δολαρίου δηλαδή. Επίσης η διάσκεψη του G20 αφορά και λίγο την προετοιμασία της Κοπενχάγης. Εσείς ε, τι βλέπετε όσον αφορά το θέμα της δέσμευσης 15-20 ε, δισεκατομμυρία ευρώ εκεί για το J20 πόσα χρήματα θα διαθέσετε. Ευχαριστώ κυρία Φόρτ. Πραγματικά ένα λεπτό παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ. Η G20 κατέληξαν σε πολλές λογικές απαντήσεις. Ότι πρέπει να επαναξεταστεί το θέμα της εποπτείας και του ελέγχου και χρειάζεται συντονισμένη προσέγγιση. Η πολιτική μας σε εθνικό επίπεδο λένε κάτι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να κάνουμε άλλα εδώ. Οι λεπτομέρειες του κανονισμού που ήδη συζητείτε από κάποιους συναδέλφους δείχνουν αποκλίσεις. και από πλευράς χρονοδιαγράμματος εκτελέσεως και όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτές καθές του κανονισμού. Οι οικονομίες μας είναι πολύ εύτραυστες. Αυξάνεται η ανεργία και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι τεράστιο πρόβλημα κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε οι Βρετανοί οι βρετανικέ ή ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να είναι σε μειονεκτούσα θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό όταν θέλουν κεφάλαιο. Πρέπει να είναι τόσο ακριβή οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να είναι σε μειονεκτούσα θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό όταν θέλουν κεφάλαιο. Πρέπει να είναι τόσο ακριβή η δανειοληψία από ευρωπαϊκέ τράπεζε, ούτω ώστε οι πελάτε, οι εταιρείε να δανείζονται από την Wall Street και να βοηθούν την Wall Street εις βάρος των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Οι εθνικοί ηγέτες υποσχέθηκαν και διακόπτεται η ομιλήτρια, κλείνει το μικροφωνό τη. Συγγνώμη, πρέπει να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Γκέρι είναι η επόμενη. Αγορήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω στα ουγγρικά. Και μπορούσα να έχω σοβαρέ συνέπειε στη Σλοβακία αν χρησιμοποιούσα αυτή τη γλώσσα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγκεκριμένοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ακολουθήσω μια. να αναφερθώ σε μια επίμαχη πτυχή τη κρίσεω. Οι Ούγγροι πολίτε εξεπλάγησαν, διότι είδαν και άκουσαν ότι οι Ουγγρικές τράπεζε. το εξάμεινο, στο, στο εξάμεινο αυτό έφτασε στα επίπεδα, στα δύο τρίτα του επίπεδου που είχαν πριν την κρίση, παρά την υποστήριξη των Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και, τρο, άλλαζαν τα συμβόλαια, τις συμβάσεις του τράπεζες και έφεραν τους καταναλωτές σε δυσχερή θέση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα στην Ευρώπη. Χρειάζεται πραγματικός έλεγχος των τραπεζών και των χρηματοστικών ιδρυμάτων διότι τα πριν που εχορηγούντο ήταν πολύ επιζήμια. Είδαμε τι αποτελέσματα έφερε. Χρειάζονται διοντολογικοί κώδικες. Να αποφευθεί η κερδοσκοπία, μακροπρόθεσμα. Χρειάζεται υπεύθυνο προβληματισμός. Ο Τσάμπα Ταμπάιτζη για ένα λεπτό. Κουρ. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής η ευρωβουλευτές μίλησαν για την ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνη των πολιτών. Να καταπολεμήσουμε του φορολογικούς παραδείσου και τα αστρονομικά πριμ. Έχω μια ερώτηση προς την Υπουργό Μάλουστρομ και τον Επίτροπο Αλμούνια. Η πρόταση του Ούγγρου Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Εποπτεία δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποια μέρα. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και των καταναλωτών που είναι εκτεθειμένοι απέναντι στις τράπεζες γιατί οι τράπεζες δεν χορηγούν επαρκή ενημέρωση για τους πολίτες. Στην Ουγγαρία ισχύει δεντολογικός κώδικας για, τους, για τις τράπεζες. Θα ήθελα να έχουμε έναν ευρωπαϊκό δεντολογικό κώδικα για να ρυθμιστεί η συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στους πολίτες. Γιατί οι πολίτες είναι τα θύματα των τραπεζών επειδή αγνοούν τους εγγενείς κινδύνους ε, στην σύναψη δανείων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, θα το εξασφαλίσουμε. Τελευταίος ομιλητής, τελευταία ομιλήτρια μάλλον στη διαδικασία του Catch the Eye είναι η κυρία Λαπάζ. Ε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, το πρόγραμμα το άκρο φιλόδοξο που μα παρουσιάσατε είναι ενδιαφέρον, αλλά μην θεωρήσετε, δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ασχοληθείτε με το κατά πόσο θα έπρεπε να ευνοηθούν οι πολύ βραχυπρόθεσμε συναλλαγέ που έχουν βραχυπρόθεσμα κέρδη και να σύγκριση να γίνει με το μεσοπρόθεσμο πρόθεσμο. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ε, προέρχεται από εκεί, από το πώς, τι γίνεται με τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Μήπως θα πρέπει αυτό το θέμα να εξεταστεί. Ε, δεν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Περίπου 8 έχω γεγραμμένου στον κατάλογο, αλλά ζητώ συγγνώμη από εσά, διότι έχουμε μόλι ένα πεντάλεπτο. Άκουσα 7, έχουμε μόνο 5 λεπτά για αυτή τη διαδικασία. Ζητώ συγγνώμη από όσου δεν είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την Υπουργό, την κυρία Μάλστρομ, να δώσει απαντήσεις. Ευχαριστώ. Θα ε, ήθελα να σας πω ότι άκουσα πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό συνένεση εδώ στην ε, Ολομέλεια για το ότι είναι σημαντικό από ευρωπαϊκή πλευρά και θα πρέπει να κάνουμε μέσα στα πλαίσια του G20. Έχουμε μια ισχυρή φωνή και συντονισμένη φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διεθνέ επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν γενικά και τον Επίτροπο Αλμούνια ειδικά που πέτυχε να οδηγηθούμε στην συνέντευξη αυτή. Αναφερθήκατε σε διάφορα από τα θέματα που θίξαμε και ο Επίτροπος και εγώ χρειαζόμαστε καλύτερο διακανονισμό των χρηματοπιστωτικών αγορών και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει το γρηγορότερα αυτό το σύστημα επιτήρησης. Αυτό προέρχεται και από την έκθεση Λεροσχέρ. Θα πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά. Χρειάζομαστε διεθνείς λύσεις πιο συντονισμένες, χρειάζομαι αποτελεσματικά μέσα σε διεθνέ επίπεδο, χρειαζόμαστε ξεκάθαρε αρχέ όσον αφορά τα συστήματα των ε, πριν και πόνου. και έχω κάθε πιστοσύνη σε, ε, ότι μπορούμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην, ε, στο 20 που θα μπορούν να συζητηθούν σοβαρά. Μετά το θέμα της χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών. Θα καλέσουμε όλες τις χώρες να τηρήσουν και να λάβουν τις ευθύνες τους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να θεωρήσουμε ότι θα συζητήσουμε για αριθμητικά στοιχεία τώρα. Αν ναι, πολύ ωραία. Χρειαζόμαστε διεθνείς λύσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ε, κοινοτικέ λύσεις κατά νου. Θα πρέπει να πετύχουμε κατά δυνατόν περισσότερες διεθνείς λύσεις. Το θέμα τώρα της ανεργίας είναι ίσως αυτό που απασχολεί τους πολίτες της Ευρώπης το περισσότερο μέσα στα πλαίσια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Γιατί η ανεργία θα παραμείνει για αρκετό χρόνο σε πολλά από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές και εθνικές λύσεις. Χρειαζόμαστε μια έντονη πολιτική για την αγορά απασχόλησης. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, να τους δώσουμε την δυνατότητα να επενδύουν και να προσλαμβάνουν. Θα πρέπει όμως βέβαια να φροντίσουμε και οι πολίτες να είναι σε θέση να απασχοληθούν καλά, να βασιστούμε δηλαδή στην παιδεία και στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση. Θα πρέπει βέβαια να μην ξεχνάμε τον Οκτώβριο υπάρχει μια ειδική συζήτηση για την ανεργία. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της πολιτικής εξόδου, γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν αρνητικές επιπτώσεις τα μέτρα που υιοθετούμε να οδηγηθούν σε ελλείμματα και σε πληθωρισμό. Και αυτό βέβαια θα πλήξει τους πιο ευάλωτους πολίτες. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε ε, και το θέμα ότι αυτή τη στιγμή στη χρηματοπιστική κρίση οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι εκείνες που το πλήττονται το περισσότερο. Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα διευκολύνουμε τους ανθρώπους αυτούς. Είναι σωστό χώρες ε, να μπορούν να βοηθηθούν από διεθνή πολυμερή μέσα χρηματοδότησης. Θα πρέπει βέβαια να φροντίσουμε να μην υπάρχει ταυτόχρονα προστατευτισμός και γι' αυτό συζητάμε διάφορους τύπους ε, διεθνούς φορολογίας όπως το φόρο και κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο διεθνώ. διεθνώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν απαραίτητε προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή και γι' αυτό θα είμαστε αντιπαραγωγικοί. Διάφοροι βουλευτές αναφερθήκαν στο θέμα των hedge funds και νέου κανονισμού στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτά είναι θέματα προτεραιότητε για τη Σουηδική Προεδρία. Είναι θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί με τους ε, ε, ευρωβουλευτές να δούμε ποιοι θα είναι οι κανόνες που θα μπορούν να ακολουθηθούν για τα hedge fund και την επιτήρησή τους. Θα υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, το ξέρω αυτό, αλλά προτιθέμεθα να συνεργαστούμε μαζί σας όσο πιο πολύ μπορούμε για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Συνοψίζοντα, κύριε Πρόεδρε, έχω να πω ότι η διάσκεψη γραφή του J20 δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα που αναφέρθηκαν εδώ. Παρ' όλα αυτά, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό βήμα προ τα εμπρό πάνω στα θέματα που εθίγησαν. Υπάρχει πίεση για τους πολίτες Ευρώπης αλλά και για όλους τους πολίτες του κόσμου. Όλοι θέλουν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να αυξήσουμε σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, να κάνουμε τα πάντα για να αποφευθούν παρόμοιες εξελίξεις στο μέλλον και να βγούμε ενδυναμωμένοι από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενωμένη είναι πολύ ισχυρή και σας εγγυώμαι ότι η Σουηδική Προεδρία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει κατά τη διάρκεια του, της G20 να προωθήσει τις ευρωπαϊκές απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Ο Επίτροπος Αλμούνια ο τελευταίος ομιλητής αυτού του θέματος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως ε, στην παρούσα συγκυρία όπου ακόμη μένεται η κρίση και έχουμε τεράστιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε παρόλο που υπάρχουν κάποια σημαντικά και αισιόδοξα μηνύματα για βελτίωση στην ανάκτηση της εμπιστοσύνη των επενδυτών στο εξωτερικό εμπόριο και η επιτυχία της Συνόδου G20 στο Πίτσμπουργκ. Και μια αξιοπιστία που θα δημιουργηθεί από την έναρξη της εφαρμογής των λύσεων στα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Γι' αυτό και όλα τα σημεία του προγράμματος εργασιών της Συνόδου Κορυφής θα πρέπει να συμφωνηθούν από τους αρχικούς κρατών και κυβερνήσεων. Και όχι μόνο να συμφωνηθούν, αλλά και να εφαρμοστούν μετά την ε, σύνοδο της επόμενης εβδομάδας. Μιλήσατε όλοι για την ανάγκη ενός απερίφραστου μηνύματος ότι οι σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου θέλουν ε, να προχωρούμε συντονισμένες δράσεις και το επόμενο βήμα στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής είναι ο καθορισμός μιας ε, στρατηγικής διεξόδου και ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για τη συντονισμένη εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Νομίζω ότι διδαχθήκαμε από το πάθημα της κρίσης ότι της κρίσης του 1929 ότι δεν θα πρέπει τα ενάυσματα να καταργηθούν πρόωρα γιατί δεν θα πρέπει να αφαιρέσουμε τα δεκαενίκια από τον άρρωστο αλλά ούτε θα πρέπει να διονυστούν αυτά τα ενάυσματα για να μην ε, επαναληφθούν οι συνθήκες που δημιουργούσαν στις πομφόλικες ε, και στις ανισορροπίες που προκάλεσαν την κρίση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να διευκρινιστούν από τη διάσκεψη κορυφής ε, του Πίτσμπουργκ. Θα πρέπει να αποφευθούν τα σφάλματα του παρελθόντο, όχι μόνο για τι μακροοικονομικέ πολιτικέ, αλλά και για τα θέματα ρυθμίση και χρηματοπιστωτική εποπτεία και δημοσιονομική εποπτεία. Αυτό φάνηκε στι προηγούμενε συνόδου κορυφή. Αναλύθη σχετική δέσμευση. Τώρα θα πρέπει να τηρηθούν αυτέ οι υποσχέσει και σε ευρωπαϊκή κλίμακα αλλά και σε παγκόσμια. Πάντως ε, συμφωνώ με όσους είπαν στην πρωινή συζήτηση ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα των πριμ. Συμφωνώ πάντως ότι το θέμα των πριμ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το θέμα των αμοιβών είναι πολύ σημαντικό και από οικονομική άποψη και από κοινωνική και από διοντολογική, ηθική και από πολιτική. Γιατί και η Ευρώπη, όπως και με άλλα θέματα του προγράμματος ε, της Συνόδου Κορυφής, ε, ανέλαβε ηγετικό ρόλο, όπως φαίνεται και από τις θέσεις των αρχηγών κρατών, αλλά και από τις θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προεδρίας. Μην ξεχνάτε ότι φέτος τον Απρίλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε στείλει συστάσεις προς τις χώρες μέλη για τις αμοιβέ. Οι συστάσεις αυτές ευθυγραμμίζονται με τις κοινώς πλέον αποδεκτές προτάσεις από όλους δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Περισσότερο κεφάλαιο, αναδιαρθρώσεις, εξηγιάνσει των τραπεζικών ισολογισμών, όχι μόνο σε ευρωπαϊκή αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Γιατί υπάρχει ε, διασύνδεση του συστήματος μεταξύ των διαφόρων συνιστοσών. Δεν μπορούμε απομονωμένα να, να προσφέρουμε κάποιες λύσεις. Γιατί μία μέρα πριν την κατάρρευση των Lehman Brothers, εμείς πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τα προβλήματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον ΗΠΑ. Αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο εξαιτία της ε, διασύνδεσης που υπάρχει. Άλλωστε, ο πολιτικός στόχος δεν είναι να εξηγενθεί ε, ο ισολογισμός μιας τράπεζας ή να κεφαλοποιηθεί το παθητικό της. Το ουσιώδες πρόβλημα έγκυται στην ανεργία, στην κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ανάγκη βιωσιμότητας και εφορίας των συστημάτων κοινωνικής μας προστασίας. Αλλά χωρίς ε, ένα εύρυθμο χρηματοπιστωτικό σύστημα όλα τα υπόλοιπα θα είναι επίσης αβίωτα και ανέφικτα. Και αυτή είναι η μείζον πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η Σύνοδος Κορυφής ε, του Πίτσμπουργκ. Μια πρόκληση που δεν είναι καινούρια. Τέλος, ε, ένα σχόλιο για κάτι που ανέφεραν πολλοί. Συμφωνώ με τα διάφορα σημεία του προγράμματος εργασιών του G20. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στους φορολογικούς παραδείσους. Η G20 δεν βρήκε λύση για όλα τα προβλήματα των φορολογικών παραδείσων. Θα ήταν δύσκολο μέσα σε μία μέρα να βρεθούν όλες οι λύσεις για ένα πρόβλημα που μας ταλανίζει χρόνια ολόκληρα. Αλλά στη διάσκεψη κορυφής, από τη διάσκεψη κορυφή του Απρίλιο μέχρι σήμερα, μέσα σε ένα εξάμεινο, έγιναν για την επίλυση αυτού του προβλήματο και για την ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών, προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και να αποκρύπτονται από τι αρμόδιε αρχέ κάποιε οικονομικέ δραστηριότητε με τη χρήση των φορολογικών παραδείσων, μέσα σε ένα εξάμεινο, επαναλαμβάνω, έγινε για το πρόβλημα αυτό πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, χρόνια ολόκληρα προηγουμένω, πριν την διάσκεψη κορυφή στο Λονδίνο. Βέβαια, μέσα σε ένα εξάμεινο δεν μπορούν να γίνουν θαύματα. Αλλά τουλάχιστον μέσα σε ένα εξάμεινο καταφέραμε πάρα πολλά για ένα πολύ σημαντικό θέμα, ώστε να αποφύγουμε κάποιε ε, δραστηριότητε που διαφεύγουν του κρατικού ελέγχου να δημιουργούν στρέβλωση στο σύστημα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε προ του Ευρωπαίου πολίτε ό,τι αφορά την ε, κατανομή του βάρους και των απαραίτητων προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τέλος, είπε κάποιος ότι η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ακούγεται πιο δυνατά από τη φωνή των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο G20. Και μέσω της Σουηδικής Προεδρίας και μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα φροντίσουμε να ακουστεί στεντόρια η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τύχει σεβασμού και προσοχής γιατί σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο μία-δύο ευρωπαϊκές χώρες ήταν αυτή που έδωσε το έναυσμα στη διαδικασία συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πιστεύουμε ότι μόνο με πραγματικό και γνήσιο συντονισμό θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την πρώτη σύνοδό μας του Οκτωβρίου. Επόμενο σημείο είναι η δήλωση του Συμβουλίου για το SWIFT και θα ήθελα ζητήσω από την κυρία Μπέτ